Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέρασε και το ακαδημαϊκό τέταρτο, οπότε δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε κι άλλο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε συνεδρίαση και το πρωί και το απόγευμα σήμερα. Συνεχίζουμε την εξέταση των σημείων της ημερήσιας διάταξης. Ε, πρώτο σημείο στην πρωινή σημερινή ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση, η γνωμοδότηση μάλλον, του κυρίου Γιάνν Χόιτεμα για την οποία έχουν κατατεθεί 515 τροπολογίες. Πληθώρα τροπολογιών, όπως βλέπετε. Αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι η Επιτροπή ΕΜΚΟ εσωτερική αγορά, αλλά η δική μας επιτροπή και η ΕΜΒΗ, δυνάμει του άρθρου 54, είναι συνδεδεμένε επιτροπές. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα συντάξει απλή γνωμοδότηση δυνάμει του άρθρου 53. Θα περάσουμε στις λεπτομέρειες με την παρουσίαση του εισηγητού του κυρίου Χαίτεμα. Παρακαλώ κύριε Χαίτεμα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, εμείς ε, με βάση το άρθρο 54 έχουμε κάποιες κοινέ αρμοδιότητες με την αρμόδια κατουσίαν επιτροπή την ΙΜΚΟ. Δυστυχώς δεν έχουμε πλήρη αρμοδιότητα για μερικά παραρτήματα που αφορούν τους ρήπους ε, από τα λοιπάσματα ή από τα προϊόντα λίπανσης. Ε, δώσαμε μεγάλη μάχη για να διεκδικήσουμε πλήρη αρμοδιότητα και για τις ρηπογόνες ουσίες. Δυστυχώς τη ε, χάσαμε αυτή την αρμοδιότητα και η ΕΜΒΗ έχει την πλήρη αρμοδιότητα για τις ρηπογόνες ουσίες των προϊόντων λίπανσης. Και το λέω γιατί έχουμε τροπολογίες σχετικές σε αυτή τη γνωμοδότηση. Πάντως ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αμερικές από αυτές είναι μη παραδεκτές, ειδικά αυτές που αφορούν τα παραρτήματα για, τα, για τις ρηπογόνες ουσίες, γιατί επαναλαμβάνω δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, πλήρη αρμοδιότητα για τα παραρτήματα για τις ρηποαντικές ουσίες ε, ε, ανήκουν στην Εύη. Οπότε οι μη παραδεκτές τροπολογίες δεν θα ψηφιστούν καν εδώ. Όσες είναι παραδεκτές θα μεταβιβαστούν στις αρμόδιες επιτροπές ΙΜΚΟ και ΕΜΒΗ για να ληφθούν υπόψη. Τώρα, ως προς τη διαδικασία αυτά, χθε, ε, σε οι για να εξετάσουν τις υπόλοιπες τροπολογίες που είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Βέβαια το θέμα αυτό είναι πολύ τεχνικό, αυτό είναι το πρόβλημα και είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες λόγω τεχνικού χαρακτήρα. Ε, του ζητήματος. Καταλήξαμε παρόλα αυτά σε νέες συμβαστικές τροπολογίες και στην πράσινη εβδομάδα μετά το Πάσχα θα επεξεργαστούμε και άλλες ε, συμβαστικές τροπολογίες. Μία πολύ σημαντική συμβαστική τροπολογία είναι για τα λοιπάσματα βραδίας απελευθέρωσης που είναι πολύ καινοτόμες ουσίες, πολύ καινοτόμα προϊόντα λίπανσης. Επίσης προσπαθούμε να βρούμε τα ελάχιστα προϊόντα θρεπτικών ουσιών στα προϊόντα λίπασης. Ε, αυτή είναι η δεύτερη συμβαστική τροπολογία. Και τρίτη, ίσως ε, καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω το δυναμικό της ε, κυκλικής οικονομίας, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο θρεπτικές ουσίες από ζωική κόπρο και όχι από ανόργανα λιπάσματα, περιορίζοντας έτσι τη χρήση των ανόργανων λιπασμάτων. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό εκεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα επίσης με τους ορισμούς και το συνδυασμό με την οδηγία για τα ζωτούχα λοιπάσματα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ο κανονισμός για τα προϊόντα λίπανσης ε, έχει κάποια σημεία που άπτονται και άλλων νομοθετικών πράξεων. Θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός γιατί υπάρχει κάποια σύγκρουση ε, αντίφαση με κάποια στοιχεία της οδηγίας για τα ζωτούχα λοιπάσματα Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε και να τα ευθυγραμμίσουμε. Ευχαριστώ και περιμένω ανυπόμονα τα σχόλια των συναδέλφων. Σας ευχαριστούμε κύριε Χαϊταμα. Ναι, ναι, ξέρουμε ποια είναι η θέση της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Βέβαια, στην Επιτροπή αυτή είναι μέλη και πολλοί ευρωβουλευτέ της δικής μας Επιτροπής, Επιτροπής Γεωργίας και παράλληλα παρακολουθούν και τις δύο επιτροπές. Αλλά φυσικά για τις τροπολογίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρμοδιότητές μας. Και σίγουρα ε, η κρατούσα θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπέρ περισσότερο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής έμβηκε για το θέμα αυτό και όχι της δικής μας. Το δικό μας ε, ζήτημα είναι η περισσότερη ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Και οι προδιαγραφές ε, που θα ε, εφαρμόσουμε για τα εισαγόμενα προϊόντα λίπανσης. Ας περάσουμε στη συζήτηση τώρα. Ζήτησαν το λόγο ο κύριος Άγνιου και άλλοι. Κύριε Άγνιου, παρακαλώ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, κυρία Αγγιλέρα. Ε, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο εισηγητής μας, ο κύριος Χαϊτεμα, είναι πραγματικά κρίμα, μεγάλο κρίμα, που δεν έχουμε την πλήρη αρμοδιότητα για τα παραρτήματα. Τελικά, η Επιτροπή Γεωργίας, σε ένα τόσο σημαντικό κανονισμό όπως είναι αυτός για τα προϊόντα ελίπασης, θα έχει ελάχιστο ρόλο, ελάχιστες δυνατότητες Τις περισσότερες αρμοδιότητες θα τις έχουν η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, για κάποιες πτυχές ακόμη και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και εμείς έχουμε σχετικά παραγωνιστεί. Όπως είπατε Πρόεδρε, φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, να ενστερνίσετε περισσότερο τη γνώμη της Επιτροπής ΕΒΗ παρά της Επιτροπής Άγκρη. Πάντω, μέσω τη συμμετοχή μα και σε άλλε επιτροπέ, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τι απόψει και τη Επιτροπή Γεωργία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χαϊτεμα όχι μόνο για τη γνωμοδότησή του, αλλά και για το συνεργατικό του πνεύμα και τη διαλλακτικότητά του και την προθυμία του για διάλογο. Χθε είχαμε, όπω είπατε, την συνεδρία στο σχεδόν εισηγητών. Είχαμε μάλιστα και την ευκαιρία να επισκεφθούμε τις κάτω χώρες και να δούμε νέες τεχνολογίες για τα όργανα λιπάσματα και τα οργανικά λιπάσματα, να δούμε τι πρόοδοση έχει σημειώσει η Ολλανδία στο θέμα αυτό, γιατί σίγουρα το μέλλον του ανήκει. Βέβαια, έχω κάποιες αμφιβολίες ε, περισσότερες από το κύριο Χαϊταμά για το κατά πόσο μπορούμε να αφιερώσουμε ε, γεωπονική μεγάλη ικανότητα στα οργανικά λιπάσματα. Γιατί ναι, μεν έχει προχωρήσει η τεχνολογία, αλλά δεν είναι τόσο προηγμένη ώστε να διαθέτουμε οργανικά λιπάσματα που θα έχουν τις ίδιες γεωπονικές ιδιότητες και ικανότητες με τα ανόργανα και που θα ανταγωνίζονται άλλα είδη λιπασμάτων όπως είναι τα ανόργανα, ή τα συνθετικά λοιπάσματα. Δεν έχουμε ακόμη προχωρήσει τόσο στην τεχνολογία στα οργανικά λοιπάσματα για να ε, παραγωνίσουμε τα ανόργανα. Πάντως, όπως είπατε, είναι πολύ τεχνικό το θέμα και γι' αυτό ήταν και πολύ δύσκολη ενασχόληση με αυτό. Χρειάστηκε μεγάλος κόπος ε, για να το παρακολουθήσουμε και ευχαριστώ θερμά τους βοηθούς συνεργάτες μου, τη Μαγδαλένα, για τη μεγάλη τους τεχνική υποστήριξη μας επέτρεψαν να εξοικειωθούμε με τόσο τεχνικές έννοιες. Έπρεπε όμως να γίνει αυτό για να μπορέσουμε να λάβουμε περιστατωμένα τη θέση μας. Και επαναλαμβάνω, οι τροπολογίες δεν είναι ούτε 52 ούτε 53. Η ομάδα μου κατέθεσε μόνο τρεις τροπολογίες. Αυτό συμφωνήσαμε με τη γραμματεία για να αποφύγουμε να κριθούν μη παραδεκτές γιατί όπως σας είπα μερικές δεν ε, εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας. Και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι αυτές οι τροπολογίες που είναι εκτός θέματος ε, να κρυθούν μη παραδεκτές, γιατί ακόμη και αν εμείς ε, τις εγκρίνουμε δεν είναι σίγουρο ότι θα ληφθούν υπόψη. Βέβαια, εναπόκειται στο συντάκτη τη γνωμοδότηση αν θα την αποσύρει όχι. Πάντω, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι όσε αρμοδι... τροπολογίε εκπίπτουν τι αρμοδιότητε τη Επιτροπή μα θα πρέπει να κρυθούν μη παραδεκτέ αυτές οι 52-53 τροπολογίες. Πάντως οι τροπολογίες των σοσιαλιστών και οι δικές μου τροπολογίες στόχο έχουν τη διευκρίνηση κάποιων ενιών. Για μας είναι σημαντική η γεωπονική ικανότητα, τα γεωπονικά χαρακτηριστικά των λοιπασμάτων. Γιατί είναι σημαντική αυτή η γεωπονική ικανότητα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διπλή χρήση των βιοτονοτικών, που είναι και φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ε, επιπλέον βιοδιαγέρτες. Μας προβληματίζει αυτή η χρήση των βιοδιαγερτικών ουσιών ή των βιοτονοτικών ουσιών. Θα το συζητήσουμε ίσως και στο μέλλον, σε μια επόμενη συνεδρίαση. Και κάτι που είπε ο κύριος Χαϊτέμα και προβληματίζει την ομάδα μου είναι ε, αυτό ότι δεν είμαι υπέρ της ε, ε, νέας οδηγίας για τα ζωτούχα για να μειώσουμε τα επίπεδα των οργανικών λιπασμάτων. Πρόκειται για ένα τεχνικό αλλά και νομικό θέμα και δεν ξέρω με τον συγκεκριμένο κανονισμό μπορούμε να ξανανοίξουμε την οδηγία για την ιτρορύπανση για τα ζωτούχα λιπάσματα. Θα πρέπει βέβαια να εκμεταλλευτούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις ώστε αυτά τα οργανικά λοιπάσματα που σίγουρα θα είναι το μέλλον ε, των λοιπασμάτων να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα γεωπονικά τους χαρακτηριστικά, τα, τις γεωπονικές τους ικανότητες. Και σίγουρα είμαστε υπέρ της κυκλικής οικονομίας, αλλά αυτή τη στιγμή λόγω της τεχνολογικής ε, πρόοδου δεν είμαστε σε θέση να γενικεύσουμε τόσο πολύ τη χρήση των οργανικών λοιπασμάτων και δεν συμφωνώ με το να ξανανοίξουμε μέσω αυτού του κανονισμού την οδηγία για τα ζωτούχα. Όπω είπε ο εισηγητή, έχουμε καταλήξει σε αρκετέ συμβαστικέ τροπολογίε και σίγουρα θα συμφωνήσουμε και σε πολλές άλλες. Με τη γνωμοδότηση του εισηγητή κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια για τα οργανικά λιπάσματα και δίνει κυρίως αυτά έμφαση και αφήνει άλλα θέματα και από αυτή την άποψη το θέμα της οδηγίας για τα ζωτούχα θα είναι ουσιαστικό ζήτημα και από αυτού θα πρέπει να τοποθετηθούμε. Εγώ είμαι κατά, επαναλαμβάνω. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Ε, πάντως θα πρέπει να δώσουμε μάχη, κύριε Χαΐτεμα, και στην ΕΜΒΗ και στην ΝΙΜΚΟ, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό να έχουμε μεταξύ μας καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ο κύριος Γιάρ. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ ε, που μπορώ να μιλήσω και πριν από τη συζήτηση των σχεδόν εισηγητών. Έχω μία γενικότερη παράκληση, διότι ο εισηγητή μα ε, σήμερα μας επισήμανε το ουσιώδες θέμα. Πράγματι, είναι αλήθεια, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να επιμερίσουμε τις αρμοδιότητες στις διάφορε επιτροπέ. Έχω όμως την εντύπωση, και θα είμαι λίγο σκληρό, ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, χωρί ε, να λάβει υπόψη τις σε τις ε, απώλειες ε, και τις παράπλευρες κυρίως απώλειες λαμβάνει συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Έχουμε δύο επιτροπές των οποίων οι πελατείες εισαγωγικά πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Όταν λοιπόν αποφασίζουμε κάτι όπου ε, τα λοιπάσματα γίνονται πιο ακριβά η οικονομία της αγοράς προφανώς και αντιδρά πάντα όταν υπάρχει έλλειψη αυξάνονται οι τιμές. Αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη όπως επίσης και οι εμπορευματικέ διαδικασίες και αυτό θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες στο εσωτερικό εμπόριο. Κατόπιν τούτου, αν θελήσουμε να ορίσουμε πολύ ψηλές οριακές τιμές, θα παρεμποδίσουμε τι αγωγέ από την Αφρική. Και διερωτώ με, ε, τι είδου αναπτυξιακή πολιτική είναι αυτή. Μα κάτι πρέπει να προσφέρουμε και σε αυτέ τι χώρε. Ε, και θα πρέπει να πω στον πρόεδρο ότι, κοιτάξτε, θα πρέπει να καλέσετε του τρει προέδρου των επιτροπών και να πούνε, ναι, πράγματι, εδώ υφίσταται πρόβλημα αυτή τη στιγμή οι επιτροπές λειτουργούν τελείως διαφορετικά, τελείως διαφορετική άποψη. Εγώ δεν έχω και αντίρρηση, αν θέλετε, όμως εγώ είμαι της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, και προσωπώ τα δικά μου σα συμφέροντα. Πρέπει όμως κανείς να στρέφει το βλέμμα δεξιά και αριστερά να δει τι κάνουν οι άλλες επιτροπές. Αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα η εξέλιξη των ε, οριακών τιμών, γιατί αυτό συζητάμε εμείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να είναι αποδεκτή για το εμπόριο και για ε, οποιασδήποτε άλλε συνέπειε μπορούν να προκύψουν. Ο στόχο δεν είναι κακό, αλλά θα πρέπει κανεί να λαμβάνει υπόψη αυτό που σα είπα και προηγουμένω παράπλευρε απώλειε. Παραδείγματο χάρη, ακόμα και οι επαγγελματικέ ε, ενώσει ε, και αυτέ αντέδρασαν γιατί υπάρχει το πρόβλημα του περίφημου limestone στα αγγλικά, ένα είδο ασβεστίου. Ε, υπάρχουν λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρες αποθήκες ε, ασβεστίου. Έτσι είναι τα πράγματα. Ε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Ως εκ τούτου, αν ληφθεί αυτή η απόφαση, θα πρέπει να κλείσουν αυτές οι αποθήκες και ο έμπορος θα είναι αναγκασμένος να πηγαίνει στη Ρωσία για να εισάγει το ασβέστιο που χρειάζεται και να μην καταφεύγει στις δικές του τις αποθήκες. Εμείς λοιπόν αν δεν ε, διατυπώσουμε αυτές τις προτάσεις μας θα γνωριτούμε. και γι' αυτό λοιπόν για άλλη μια φορά παρακαλώ οι τρεις άμεσα εμπλεκόμενοι πρόεδροι επιτροπών να ξανασαντηθούν και να πούν ότι πράγματι έχουμε λάβει υπόψη μας ε, όλα αυτά τα οποία θα προκληθούν από τις αποφάσεις μας. Γιατί ξέρετε, δεν πρόκειται μόνο για ένα τεχνικής φύσεως θέμα. Διακυβεύονται πολλά περισσότερα και αυτή τη στιγμή σας λέω και πάλι οι επιτροπές ακολουθούν τελείως διαφορετική κατεύθυνση στην Ολομέλεια. Είμαστε και ειλικρινεί εκεί. Μερικέ ε, φορέ οι ψηφορίε είναι τυχαίε, εξαρτάται από το τι διάθεση έχει κανεί, πώ έχει ξυπνήσει. Το λέω τώρα για πολλωστή φορά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει πράγματι ο πρόεδρο να συγκαλέσει του τρει πρόεδρους επιτροπών για να συζητήσουν για το θέμα. Κοιτάξτε, το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε στο τέλο, ε, κανεί να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερα. Αυτή τη στιγμή βλέπω βλέπω να υπάρχουν πολλές, ε, πολλοί φόβοι ότι, όπως σας είπα, θα αυξηθούν οι τιμές και θα περιστούν και οι εμπορικές σχέσεις. Και τελευταία μου παρατήρηση σε αυτά που είπε ο εισηγητής για τα οργανικά λοιπάσματα. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ καλή συμφωνία ε, διότι οι γεωργοί ε, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες με τα οργανικά λιπάσματα και δεν μπορούν εύκολα να τα χρησιμοποιήσουν γιατί οι νόμοι είναι όλο και πιο σκληροί. Εγώ λοιπόν θα θεωρούσα σωστό ε, να πούμε ότι κοιτάξτε από πλευράς νομοθετικής δεν υπάρχει μόνο ένας άκαμπτος νόμος αλλά μπορούμε να βρούμε και μία άλλη λύση δηλαδή να μπορεί κανείς τα οργανικά λιπάσματα να τα τροποποιήσει, να τα μεταποιήσει. Αν η τεχνολογία υπάρχει, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή προσφορά ε, προς τους γεωργούς. Όχι δηλαδή να τους λέμε, ξέρετε αυτό είναι και δεν υπάρχει λύση, όχι να τους πούμε ότι ξέρετε έχουμε και κάποια εναλλακτική λύση. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους προελίσσαντες. Ξέρουμε πόσο απαιτητικό είναι αυτό το νομοθέτημα και από τεχνικής πλευράς και γεωπολιτικής αλλά και για ιδεολογικούς λόγους. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ε, γι' αυτό το λόγο, μεταξύ άλλων, κατά τη σύνταξη αυτή του νομοθετήματος ε, συγκαλέσαμε τόσες ε, τεχνικές συνεδριάσεις για να παρουσιαστούν οι διάφορες απόψεις. Αν δούμε τώρα τα πορίσματα, διαπιστώνουμε πως η αρχική πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κάδμιο, για τα φωσφορούχα, για, κάποιες, ε, ε, για κάποιους τομείς απεδείχθη υπερβολικά φιλόδοξη. Ε, και προσπαθούμε να έχουμε αυστηρότερε οριακέ τιμέ κατά τρεις ή τέσσερις φορές ε, αν, αν συγκρίνουμε την κατάσταση με αυτή που επικρατεί σε άλλες χώρες. Επίσης, οι ειδικοί στον τομέα της υγείας είχαν την ίδια άποψη. Δεν θεωρούν ότι πρέπει να μειώσουμε τόσο πολύ τα επίπεδα καθμίου. Όχι ότι αυτό είναι αρμοδιότητά μας, ε, αλλά είναι και προς συμφέρον μας. Η κυρία Καμπίνη που είναι η συγγήτρια για την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, παρουσίασε αυτά τα ζητήματα. Δύσκολα μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με οικοδομητικό τρόπο αν ακολουθηθεί τελικά αυτή η κατεύθυνση. Για την έκθεση του Γιάννου, θέλω να σε ευχαριστήσω για την ημερίδα μελέτης στην Ολλανδία Νομίζω ότι είναι η σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ε, θα πρέπει η ζωική κόπρος να έχει ιδιαίτερο καθεστώς για τη χρήση της στα οργανικά λοιπάσματα. Νομίζω ότι πρέπει να προωθήσουμε ε, την ε, κατεύθυνση αυτή, διότι για την κυκλική οικονομία, αν έχει μια ευκαιρία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η γεωργία, λοιπόν αυτή είναι. Δηλαδή η χρήση των οργανικών λοιπασμάτων. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε τα ποσοστά. Όμως, ε, διαπιστώνουμε ότι η Ψαλίδη είναι ευρεία και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ε, το ζήτημα είναι να βρίσκουμε τεχνικά εφικτές λύσεις ε, και αυτό προτείνεται στη γνωμάτωση του Γιάννη. Ε, για το πόσο είναι αποδεκτή κοινωνικά η γεωργική πολιτική. Ο κύριος Γιάρ μα είπε χθε πως ε, λόγω του, της πολιτικής ατμόσφαιρας είναι σχεδόν απαράδεκτη η, η χρήση των λοιπασμάτων και ότι δεν γίνεται, μας είπατε δεν γίνονται αντιληπτές ε, οι αρνητικές συνέπειες της απόφασής μας. Βεβαίως, θα πρέπει να δούμε πώς βλέπουν οι άνθρωποι τις αποφάσεις μας. Ε, δηλαδή, να προσπαθήσουμε να αντιπροτείνουμε λύσεις τύπου κυκλικής οικονομίας. Η νητρορύπανση, οι οδηγίες για τα ζωτούχα ε, θα ε, δημιουργήσουν πολλά προβλήματα αν τις διαπραγματευτούμε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Μόνο και μόνο ο τίτλος τροποποιούμε τον κανονισμό για τα ζωτούχα και ε, την ε, περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία των οργανικών λιπασμάτων, όπως φαίνεται από τον τίτλο. Νομίζω πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα λιπαντικά αποτελέσματα των οργανικών λιπασμάτων και τις λιπές συνέπειες αυτών των ουσιών, ούτως ώστε να είναι ε, καλά ε, στοιχειοθετημένη η θέση που θα υπερασπιστούμε και να βρούμε ε, πρόσφορες λύσεις ούτως ώστε να είναι αποδεκτή η λύση που θα βρούμε και από τους γεωργούς. 800 τροπολογίες από την Εύη. Συνολικά καταλήξαμε σε 500 τροπολογίες. Ελπίζω πραγματικά να μην βαρύνουμε τη γεωργική πολιτική με αυτά που θα αποφασίσουμε και να βρούμε μια γενικά αποδεκτή λύση. Ευχαριστούμε, Άντριο. Αντρία... Άγνιο, συγγνώμη. Πίτερ, θα αναφερθώ σε σένα, άκουσε με τι λέω. Ένα λεπτό να κάτσει ο κύριος Γιάρ, γιατί θα μιλήσω για αυτόν. εξεπλάγει και δεν δυσκολεύομαι να πιστέψω, πιστέψω αυτά που άκουγαν τα αυτιά μου όταν μιλούσε ο Πίτερ Γιάρ. Μας μιλάει για τη, τα αποθέματα καδμίου και για τον ασφαιστόλιθο. Αυτά μόνο σας προβληματίζουν για την γεωργική γη. Ε, και λέτε ότι δεν θα έχουμε αρκετά και πρέπει να τα εισάγουμε από τη Ρωσία. Μα Ελπίζω η Επιτροπή να ξέρει ότι όταν χρησιμοποιούμε ασβεστόλιθο για τη γη, τόνους ολόκληρους χρησιμοποιούμε ένα εκτάριο πελώριες ποσότητες και είναι ξερό υλικό, έτσι, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Το κόστος είναι, τι να σας πω, εξωφρενικό για εισαγωγή από τη Ρωσία. κανέν μας δεν μου το είχε πει αυτό από τους Γεωργούς και ε, δεν ξέρω, ε, μήπως ανακάλυψες εσύ κάτι και πρέπει να μας διαφωτίσεις όλους. Αλλά πάντως όσοι είναι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ε, θα πρέπει ίσως να συνειδητοποιήσουν αυτό το, αυτό μήνυμα και ο Μάρτιν Χόισλινγκ νομίζω θα με υποστηρίξει διότι ε, και για την βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί το ασβεστόλες και δεν νομίζω να ε, τους δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ας έχουμε ένα κοινό γεωργικό μέτωπο και ας κάνουμε κάτι γιατί αλλιώς θα περάσει τα ψηλά τα γράμματα και τότε θα έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα. Τώρα ο κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ. Διαπιστώνεται και από τι παρατηρήσει και τα σχόλια ότι είναι πολύ σύνθετο και περίπλοκο το θέμα, όχι μόνο γιατί είναι τεχνικό περίπλοκο, αλλά γιατί έχει και μια έντονη πολιτική διάσταση και δεν είναι τυχαίο που εμπλέκονται εδώ όχι τρει αλλά τέσσερι επιτροπέ. Ε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος γιατί έχει ε, περιβαλλοντικές συνέπειες, ε, η εσωτερική αγοράς, εμείς φυσικά, αλλά και ακόμη και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εξού και η ιδιαιτερότητα αυτού του θέματος με την εμπλοκή τόσων πολλών επιτροπών. Και ευχαριστώ τον κύριο Χαίτεμα για το έργο του, για τις προτάσεις που μας υπέβαλε. Και όπως είπε και η κυρία Αγγιλέρα, και εγώ έχω πολλές απορίες και προβληματισμούς, αλλά περιμένω τις συγκεκριμένες συμβαστικές προτάσεις για να αποφανθώ. Πάντως πιστεύω θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά την ε, αμφισβήτηση ή την επανάληψη της συζήτησης για την οδηγίες για την νητρορύπανση. Και συμφωνώ με πολλές προτάσεις για τα λοιπάσματα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να είμαστε σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά την επεξεργασία της ζωικής κόπρου επιτόπου. Ναι, είμαι υπέρ της κυκλικής οικονομίας, αλλά προσοχή να, μην παράγουμε επιτόπου ένα λοιπάσμα με τη λογική να το μεταφέρουμε σε μεγάλες αποστάσεις. Δεν μπορούν αυτά τα προϊόντα να χρησιμοποιούνται μακριά από τον τόπο παραγωγής οπότε έτσι να χάνουμε ε, τα πλεονέκτηματα της κυκλικής οικονομίας ε, λόγω της μεταφοράς σε μεγάλη διάστα... Ε, απόσταση και την μεγάλη απόσταση που χωρίζει τον τόπο παραγωγής από τον τόπο χρησιμοποίησης. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα κόστος, γιατί μπορεί να επηρεάσει την οικονομία της γεωργικής εκμετάλλευσης σε ένα υπερβολικό κόστος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντελαέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χαϊτεμα για το έργο του, πολύ αξιόλογο. Εγώ επειδή είμαι γεωργός και χρησιμοποιώ φυσικά λιπάσματα, είτε χημικά είτε οργανικά, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να κρατήσουμε τον κοινό νου σε τέτοια θέματα και έχουμε την αίσθηση ότι όταν ε, παρακολουθούμε τις συνεδρίες εμείς επιτροπής έχουμε μια θέση και μετά σε άλλη επιτροπή έχουμε άλλη θέση. Εδώ εμπλέκονται πολλές επιτροπές όπως είπαμε. Και μερικές φορές επιφορτίζουν τους συναδέλφους τους ε, στη μία επιτροπή να πείσουν τους άλλους συναδέλφους ε, σε άλλη επιτροπή που επίσης εμπλέκεται στο θέμα. Και άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Αντριέ και τα λαμβάνω υπόψη, αλλά το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Η ιδανική λύση δεν υπάρχει το μη χειροβέλτιστο θα μπορούσαμε να πούμε και από τη στιγμή που ε, θέλουμε την κυκλική οικονομία θα πρέπει ε, η ζωική κόπρος των ζώων που θέλουμε να καταναλώσουμε να μπορούν να αξιοποιούνται στη γεωργία. Το καλύτερο φυσικά θα ήταν να χρησιμοποιείται όσο πιο κοντά στην παραγωγή γίνεται αυτή η ζωική κόπρος. Αλλά δεν μπορούμε σε ένα νομοθετικό κείμενο να υποχρεώσουμε την κατανάλωση επιτόπου, τη χρησιμοποίηση επιτόπου ε, τέτοιων λοιπασμάτων. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς λοιπόν και εμείς που εδώ ε, υπερασπίζουμε την γεωργία και την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή θα πρέπει να πείσουμε τους συναδέλφους σε άλλες επιτροπές περιβάλλοντος, διεθνούς εμπορίου, εσωτερικής αγοράς να λάβουν υπόψη την γνώμη της Επιτροπής Γεωργίας γιατί είμαστε ενία και αδιέρετοι. Ευχαριστώ πολύ συχνά μας ε, μένφονται ότι είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι, γιατί είμαστε πολύ κοντά στους γεωργούς. Ε, οι περισσότεροι από μας είμαστε και αγρότες, ε, έχουμε γεωργική παραγωγή. Α, αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να στερηθούμε τις αρμοδιότητες σε αυτό το θέμα. θα πρέπει να μπορούμε και εμείς να επηρεάσουμε την όλη συζήτηση. Κυρία Μακίνταερ. Uh, Um... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους ε, προλαλήσαντες ότι πράγματι υπάρχουν σε αυτή την Επιτροπή πάρα πολλοί γεωργοί, καλλιεργητές και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί η φωνή της ε, γεωργίας. Εναπόκειται λοιπόν σε εμά ε, να υπερασπιστούμε τους γεωργούς σε ολόκληρη την Ευρώπη οι οποίοι απελπισμένα ζητάνε την πρόσβαση σε λοιπάσματα μεταξύ βέβαια και άλλων προϊόντων και σε άλλα προϊόντα. Ανησυχούμε για την ασφάλεια των τροφίμων, για την ε, αυξανόμενη παραγωγή. Προφανώς και πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία των λιπασμάτων. Όπως και πολλοί άλλοι προλαλήσαντες ε, σήμερα το πρωί και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για το ότι οι αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής ε, περικόπηκαν ουσιαστικά και θέματα όπως το κάδμιο, το οποίο είναι πολύ επίμαχο και όπου νομίζω ότι οι προτάσεις της Επιτροπής είναι πολύ προχωρημένες. Σε τέτοιου είδους τομείς θα ήθελα να έχουμε αρμοδιότητες. Παρ' όλα αυτά ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του και για το ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ε, γεωργίας. Εγώ έχω καταθέσει μία σειρά τροπολογιών. Ε, δεν θα προσπαθήσω να επαναλάβω αυτά που ελέγχθησαν. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που ελέγχθησαν. Νομίζω ότι τελικά σε οποιαδήποτε νομοθετική πράξη προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου το διοικητικό βάρος το οποίο επιβάλλουμε στους ανθρώπους, είτε είναι οι ίδιοι γεωργοί, είτε αν θέλετε στους ε, παραγωγούς ε, λιπασμάτων στην περίπτωσή μας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ένα είδος ε, λογικής, ένας κοινό νους να χαρακτηρίζει τις προτάσεις μας. Παράδειγμα, η δική μου τροπολογία στο παράτημα 4 τμήμα 2.2 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον σχεδιασμό ε, προγράμματα όπου εντοπίζονται συγκεκριμένοι τομείς. Εγώ στη μέση βλέπω ότι πρέπει να υπάρχει ε, και ένα διάγραμμα της διαδικασίας παραγωγής, συγκεκριμένα γραπτή περιγραφή της διαδικασίας. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό. Μα αυτό δεν είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του προϊόντος. Ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί σε αυτά που ε, περιλαμβάνονται σε νομοθετικές πράξεις και στις επιπτώσεις ε, που απορρέουν, πρόκειται για την αύξηση του διοικητικού βάρους. Καταλαβαίνετε, <clears throat> αυτό είναι και επίθεση στον ανταγωνισμό, επίθεση έναντι των επιχειρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να διασφαλίσουμε στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τη θέση των γεωργών, ε, των καλλιεργητών, αλλά επίσης ε, και να λάβουμε υπόψη μας την ανάγκη να υπάρχει καλύτερη να υπάρχουν καλύτερε νομοθετικέ ρυθμίσει. Μιλάμε πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Νομίζω πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε περνάει από εδώ ως απόφαση θα πρέπει να καλύπτει αυτές τις προδιαγραφές της ε, καλύτερης νομοθετικής διαδικασίας και θα εξετάζει τις επιπτώσεις των νομοθετικών πράξεων κυρίως εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Όντως δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο το θέμα αυτό και έχει και πολλές διακλαδώσεις εξού και η πολυπλοκότητά του. Φυσικά ε, θέλουμε μείωση της χρήσης των λιπασμάτων, ε, διατηρώντας όμως υψηλή ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, ε, με σεβασμό της, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας καθώς και της υγείας των ζώων. Και υπάρχουν κάποιες αλληλεπιδράσεις με την οδηγία για την ιτρορύπαση. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο ρόλο των βιοδιαγερτών ή βιοτονοτικών υλικών. Έχω τις τροπολογίες 80 και 188. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε αυτή την πρακτική για να ενισχύσουμε τη θρέψη των φυτών και να προστατεύσουμε τους σπόρους. Οι μικροοργανισμοί φυσιολογικής προέλευσης που ενισχύουν τη θρέψη των φυτών θα πρέπει να θεωρούνται ως βιοτονοτικά υλικά, βιοδιαγέρτες. Και μάλιστα ενισχύονται την έρευνα για τις ουσίες αυτές, αυτούς τους φυσικούς βιοδιαγέρτες, ε, νομίζω ότι θα αναπτύξουμε μία υγιεινή και ποιοτική γεωργία και θα περιορίσουμε τη χρήση των τοξικών λιπασμάτων. Νομίζω ότι αυτό θα εξυπηρετήσει και τους γεωργούς. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Περιμένουμε τον κύριο Χόισλινγκ και τι θα μας πει. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να βάλουμε και τα κλάματα που έχουμε μικτές αρμοδιότητες και οι υπόλοιπες επιτροπές θα ήθελαν περισσότερες αρμοδιότητες. Τώρα για το κάδμιο, καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχουν ανησυχίες Και όταν βλέπω πώς ήταν και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, καταλαβαίνω γιατί ανησυχούν μήπως ληφθεί αντίθετη απόφαση. Ο της ηγητή τη ομάδα μα ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντο έχει αυτή την άποψη και το καταλαβαίνω και φυσικά θα τον υποστηρίξουμε. Ε, φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, διαστάσεις της υγείας και της χρήσης υγιεινέστερων οργανικών λοιπασμάτων. Δεν μπορεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα τομέα να έχει ε, διαφορετικές επιπτώσεις από τη γενική κατεύθυνση που ακολουθούμε. 60% ε, της μόλυνσης από το κάδμιο προέρχεται από τα λοιπάσματα. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα και φυσικά πρέπει να μειωθούν οι οριακές τιμές. Τώρα καταλαβαίνω τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων κρατών μελών και τη βιομηχανία. Ξέρω δεν μπορεί να είναι υποδεέστερο ο ρόλο. Το αντελήφθην κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Δεν μπορούμε όμω. Εμεί εκπροσωπούμε εδώ τη γεωργία. Και τα χημικά λοιπάσματα ε, που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να περιοριστούν. Και όταν μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 20 γραμμάρια, δεν ξέρω καν τεχνικώς είναι εφικτό αυτό. Ε, δεν μπορούμε εμείς να υιοθετήσουμε αντίθετη άποψη και μετά τι θα κάνουμε στην Ολομέλεια. Όταν βλέπουμε ε, ότι ε, αυτοί που θα έπρεπε να υπερασπίζουν το περιβάλλον τελικά ε, υιοθετούν λύσει που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ε, για την νητρορύπανση και την οδηγία για τα ζωτούχα, Ε, ξέρω τι θα μας πούνε, ότι όλοι ε, θε, θεωρούμε ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα ε, έχουν υποδεέστερη θέση. όχι, δεν ισχύει αυτό. Ε, όταν ο Πίτερ Γιάρ θέλει να, δεν μας όλα τα άλλα, θέλει να καλύψει, να καλέσει την Επιτροπή Ανάπτυξης για να βλέπουμε και τα προβλήματα που δημιουργούμε στην Αφρικανική Ήπειρο, συγγνώμη, αλλά ε, δεν μπορούμε με σοβαρότητα να το ε, ισχυριστούμε αυτό, θα πρέπει με κάθε σοβαρότητα αντίθετα να καλέσουμε όλες τις αρμόδιες επιτροπές και να σεβαστούμε όλες τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια. Βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση ε, και με την έκθεση που αφορά τα, τα, ε, τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Και φυσικά η Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να είναι αρμόδια. Είναι δυνατόν ε, η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού να επιλαμβάνεται του τους αυτού. Εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας ε, ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. που θα μας κάνει να προσετεριστούμε και τον κλάδο. Και φυσικά θα μιλήσουμε για, για το περιορισμό του καδμίου στην Επιτροπή Γεωργίας, αλλά να μην ξεχνούμε και τις πληροφορίες που μας δίνουν οι ενδιαφερόμενοι. Η μόνη χώρα που έχει ε, λιπάσματα με τέτοια όρια καδμίου είναι η Ρωσία, μην το ξεχνάτε και ο ευρωπαϊκός κλάδος παραγωγής χημικών προϊόντων θα υποφέρει με μια τέτοια διάταξη και θα ευνοήσουμε τη ρωσική βιομηχανία. Εμείς θέλουμε μια, έναν οικολογικό κλάδο παραγωγής α, ε, λιπασμάτων, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι δύνατο να έχουμε αποτελεσματική γεωργία χωρίς χημικά λιπάσματα. Αυτό αποκλείεται. Ο κύριος Καπούτο. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του. Προφανώς δεν θα επαναλάβω όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τους συναδέλφους και δεν θα επαναλάβω αυτά που ελέγχθησαν για το κάτμιο. Όμως ε, ε, θέλω να διευκρινίσω δύο θέματα πρακτικής φύσεως ε, για τους γεωργούς, οι οποίοι όταν αγοράζουν λιπάσματα θέλουν η ποιότητα είναι αυτή που αναφέρεται στον κανονισμό. Σήμερα λοιπόν, οποτεδήποτε αγοράζουν λιπάσματα με κάδμιο, κάλιο, αζωτούχα, συνθετικές ουσίες, σε αυτή τη σύνθεση που αναφέρεται, πρέπει η ε, σύνθεση που ισχύει να τηρείται στο σύνολο των θρεπτικών ουσιών. Με την πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν αυτή τελικά περάσει, η υγειοργή ε, περίπου ένα 6%, το 2 δηλαδή θα πάει στο 6% και κατόπιν τούτου το 15-15-15 θα μπορεί να μετραπεί σε 13-13-13 στις συνθέσεις των θρεπτικών ε, ουσιών. Εγώ έχω καταθέσει μία πρόταση. Άζωτος, ε, άζωτο, φόσφορο και ποτάσιο και κάλιο, με συγχωρείτε, ε, αυτά να παραμείνουν στις σωστές αναλογίες Ας μην ξεχνάμε ότι περίπου το 5% της απόκλησης, γιατί προβλέπεται αυτή η δυνατότητα απόκλησης, ε, αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό. Οι γεωργοί θέλουν να αγοράζουν ένα τόνο, ας πούμε, ε, λιπάσματα και να μην αγοράζουν σχεδόν πολύ λιγότερο από το πραγματικό βάρος. Εξάλλου, θέλω να πω ότι οι γεωργοί επιθυμούν να έχουν την εγγύηση ότι τα λοιπάσματα θα δίδουν τις τρεπτικές ουσίες ε, που θα προσαρμόζονται στο δικό τους πολιτισμό, γιατί θέλουν να θρέψουν τα φυτά. Όσον αφορά το φόσφορο, εδώ το θέμα κλειδί για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα για τα φυτά είναι να υπάρχει μια διαλυτή ε, φόρμουλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει να φέρεται η περιεκτικότητα φωσφόρου στην ετικέτα, αλλά όχι η διαλυτότητά του. Κατόπιν τούτου, εγώ και για αυτό το θέμα κατέθεσα μία τροπολογία, έτσι ώστε να υπάρχουν τα ελάχιστα επίπεδα διαλυτότητας για τα ορυκτά λιπάσματα που αναφέρονται στο παράρτημα. Ελπίζω λοιπόν, όσον αφορά ε, αυτά τα ε, ανόργανα λοιπάσματα ε, να περάσει αυτή η τροπολογία που σας έχω καταθέσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή που μας κατέθεσε αυτήν την έκθεση ε, και θα ήθελα να πω ότι αυτές οι ορικές τιμές δεν ισχύουν γιατί ξέρουμε παρήματος χάρη στα αζωτούχα λοιπάσματα Εκεί έχουν γίνει συγκεκριμένες έρευνες και έχει διαπιστωθεί ότι μέχρι και 350 κιλά εφόσον χρησιμοποιηθούν μέχρι και 35 κιλά τελικά δεν προκύπτει η δυνατότητα να φύγουν τα λοιπάσματα αυτά σε λεκάνες αποθήκευσης υδάτων. Γι' αυτό λοιπόν δεν το βρίσκω σωστό αυτό που αναφέρεται σχετικά με τις οριακές τιμές. Προφανώς και θέλουμε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον, αλλά το να πούμε ότι ε, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση με κάδμιο, Πρόσφατα μου είπε ένας καθηγητής ότι δεν είναι έτσι ακριβώς γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου προκύπτει ουσιαστική επιβάρυνση με κάδμιο. Ε, νομίζω λοιπόν ότι όσον αφορά τώρα το θέμα της εξάρτησης από τη Ρωσία, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε κατά πόσον πρέπει να το επιτρέψουμε, δηλαδή να είμαστε εξαρτημένοι από τις επιταγές της ε, Ρωσίας. Τώρα, όσον αφορά την όξινη βροχή, καλό αυτό που τη συζητάμε, θα πρέπει όμως ε, να συζητήσουμε λιγάκι και για το θείο. Έχουν γίνει έρευνες και το αρμόδιο συστούτο διαπίστωσε ότι στο έδαφος δεν υπάρχει αρκετό θείο, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ε, χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα λιπάσματα είναι ε, απαραίτητο να υπάρχει χρήση των σωστών λοιπασμάτων αν θέλουμε πραγματικά να διατηρήσουμε την απόδοση στο επίπεδο που θα πρέπει. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ε, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, ούτε να επαναλαμβάνω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ε, κυρίως ε, ο Αντριέ, ο Ντενανό και τα λοιπά. Θα είμαι σύντομος. Ε, κάποιοι συζήτησαν το ενδεχόμενο επανεξέταση ε, τη οδηγία για τα ζωτούχα. Λοιπόν, για αυτό το θέμα υποστηρίζω πλήρω τη συνάδελφα Αγγιλέρα. Να μην το ξανανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό. Ε, δεν ε, είναι καταλληλότερη λύση για να δώσουμε ένα, ε, μια απάντηση για αυτό το ζήτημα που είναι τόσο σημαντικό για τη Γεωργία. Θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Γιατί ε, στο μέλλον ίσως ναι χρειαστεί αναθεώρηση γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία αλλά δεν θα πρέπει να την αναθεωρήσουμε χρησιμοποιώντας ως όχημα αυτή την οδηγία ή οποιαδήποτε άλλη οδηγία και θα υποστηρίξουμε και το σκιώδη μας ε, στην ΥΠΚΟ. Ο Πίτερ Γιά. Ναι. Ευχαριστώ. Για το κάδμιο δεν είμαι γεωλόγος, αλλά ε, στην Ευρώπη δύο περιοχές είναι όπου μπορούμε να βρούμε ασβεστόλιθο ε, και ε, μιλάμε για περιοκτικότητα σε διάφορα μείγματα στην ανατολική Γερμανία και στην Πολωνία. Στην περιοχή μου, παραδείγματος χάρη, Έχουμε 50 χιλιόμετρα απόσταση μέχρι το σημείο που υπάρχει ο σβεστόλιθος. Καταλαβαίνετε πόσο κοστίζει αυτό για τις μεταφορές. Ε, και για την Ευρώπη, είπα, εξαρτάται από πού προέρχεται ο ασβεστόλιθος. Ε, και όταν μιλάμε για ε, τριπλάσια οριακή τιμή, δεν είμαστε ακριβώς συγκεκριμένοι. Και ναι, κύριε Ντέσπορ, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, οι τρει αρμόδιες επιτροπές, ξαναλέω, πρέπει να συζητήσουν, να βρουν μια εξορροπημένη λύση. Δεν είναι ότι θέλουμε να επιβάλλουμε την άποψή μας, αλλά δεν θέλω στο τέλος να έρθει κάποιος και να μας πει «Α, δεν το ήξερα». Ε, καλές οι αρμοδιότητες, καλή οριοθέτηση των αρμοδιότητων μας, αλλά να μην παραπλανούμαστε. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε με κατεύθυνση ακολουθούμε. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και την διαβούλευση με τη Σνάλφο Γκαρντίνη. Έχω την εντύπωση ότι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, από τη συζήτηση προκύπτει δηλαδή ότι δεν υπάρχει κατανόηση για βασικά ζητήματα. Γι' αυτό λέω πρέπει να ανταλλάξουμε πληροφορίες με τους συναδέλφους ε, και να ε, οι συνάδελφοι από τι Επιτροπέ και οι πρόεδροι των ε, αρμοδίων επιτροπών να συζητήσουν. Ε, εγώ καταλαβαίνετε ότι δεν θέλω να πετάμε όλα τα σκουπίδια στις διπλανές αυλές. Αυτό έλεγα. ακολουθούμε μια κοινή γραμμή στην Ευρώπη και ε, δεν μπορούμε ε, να πάρουμε τις αποφάσεις όπως μας βολεύουν εμάς. Πρέπει λοιπόν να ξέρουν και οι τρεις επιτροπές ε, τι ακριβώς θα προκαλέσουν με τις δικές τους αποφάσεις. Το monitoring, αυτός ο έλεγχος που προτείνω, είναι μια, ένας διακαής πόθος μου, έτσι ώστε στο σημείο αυτό να μην υπάρχουν αποκλίνουσες στρατηγικές και πορείες. Κυρία Σλάιερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 1990 είχα λάβει μέρος σε πολλές ε, συνεδριάσεις που μιλούσαμε με τους γεωργούς για τις οριακές τιμές ε, των αζωτούχων λοιπασμάτων. Έχουμε φτάσει το 2017 και πρέπει να δούμε αν τηρούνται αυτές οι οδηγίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χαΐταμα για την εξαιρετική του έκθεση και να πω ότι ε, δεν έχουμε προχωρήσει πολύ από το 1990. Και τελικά θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις θέσεις των δύο επιτροπών, Άγκρη και Έμβη. Είμαι τακτικό μέλος και στην Επιτροπή Έμβη και πιστεύω ότι και ο ο ε, γεωργικός κλάδος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κυκλική οικονομία. Και είναι σημαντικό ε, γιατί χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία και άλλα στοιχεία, άλλα δεδομένα από αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής. Οι μη, θα κολλήσουμε. Και θα πρέπει να προστατεύσουμε και την ξηρά και το νερό και τον αέρα, την ποιότητα του αέρα. Επίσης, ε, η σημαντικό θέμα η επαναχρησιμοποίηση κάποιων πρώτων υλών. Ε, και τι ε, μας λείπουν, φωσφορικά άλατα. και τα φωσφορικά άλατα είναι χρυσάφι για τη γεωργία. Γι' αυτό και επενδύουν εκεί πολλές χώρες, όπως η Κίνα για παράδειγμα. Θα πρέπει να είμαστε, δεν πρέπει να είμαστε ε, αυστηροί και σκληροί απέναντι στους γεωργούς, γιατί και αυτοί θα πρέπει να επιβιώσουν, ιδιαίτερα οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι ε, θα επικρατήσουν παντού οι πολυεθνικές και θα απορροφήσουν τις μικρές ε, επιχειρήσεις. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είχαμε πολύ καλή συζήτηση, γιατί ακούσαμε και τη γνώμη των ενδιαφερομένων. Και φυσικά χρειαζόμαστε πόρους, κονδύλια και γιατί όχι και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία. Οι Επίτροποι Φέλερ και Χόγκαν συμφωνούν, αλλά προσκρούν στις αντιδράσεις του λόμπι των παρασκευαστών συνθετικών λοιπασμάτων, που δεν είναι μόνο στην Ρωσία και στην Ιταλία, στην Πολωνία, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν έχουμε παραγωγούς συνθετικών λιπασμάτων. Πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και τα συνθετικά λιπάσματα φυσικά χρειάζονται. Χρειαζόμαστε και οργανικά αλλά και συνθετικά λιπάσματα. Και αυτό χρειάζονται οι γεωργοί. Το γνωρίζουμε όλοι ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τέτοια συνθετικά λοιπάσματα, Γεωργή, και δεν είναι τα συνθετικά λοιπάσματα υποκατάστατο των ζωικών, των οργανικών. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Επίσης είπε ότι εκπλείονται τα συνθετικά λοιπάσματα και φτάνουν στον, ε, στον υδροφόρο ορίζοντα ε, μολύνοντας το νερό. Αλλά και με τα λοιπάσματα μπορούμε να διαχωρίσουμε το μολυσμένο νερό από το νερό που δεν έχει ρηπανθεί. Επίσης θα πρέπει να σεβαστούμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες που είναι υπερβολικά αυστηροί και θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις ε, ανόργανες που είναι πολύ χρήσιμες. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για την ε, ε, νητρορύπανση και τα ζωτούχα, Θα ήθελα να σας παραπέμψω στον ε, Ολλανδό Υφυπουργό ε, Περιβάλλοντος που έχει πολύ καλή θέση. Εμείς θέλουμε όλες αυτές τις θρεπτικές ουσίες να φτάνουν στο φυτό, να φτάνουν στο έδαφος και αυτό επιδιώκει και ο Γιώργος, αλλά δεν το καταφέρουμε εξαιτίας αυτής της οδηγίας για τα ζωτούχα, για την μητρορύπανση. Και εξού και η τραγωδία που βιώνουμε στις κάτω χώρες επειδή οι γεωργοί ε, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν όπως θα ήθελαν τα χωράφια τους εξαιτίας αυτής της οδηγίας για την ιτρορύπανση. Έχω καταθέσει πολλές τροπολογίες και εγώ γιατί πάντα καταθέτω τροπολογίες και στις διεπιτροπές και στην Επιτροπή Γεωργίας και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και φαίνεται ότι θα κρυθούν μη παραδεκτές μερικές τροπολογίες. Για το κάδμιο, για παράδειγμα, έχουμε πολύ καλές τροπολογίες ενός Γάλλου συναδέλφου και είναι απαράδεκτο να κρυθούν απαράδεκτες οι τροπολογίες αυτές. Και αν πραγματικά θέλουμε στο μέλλον ε, να, έχουμε σημαντικό ρόλο στην ε, παγκόσμια γεωργία, δεν πρέπει να περιθεροποιήσουμε τους γεωργούς μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οριακέ τιμέ που θα θεσπίσουμε θα πρέπει να είναι ρεαλιστικέ για να μπορέσουν να τι σεβαστούν οι γεωργοί, να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να μην, να μην οδηγηθούν σε αφανισμό. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας. Ε, να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα για την ε, μεικτή αρμοδιότητα. Προσοχή. Όλες τις αντίστοιχες επιτροπές μας ε, θα πρέπει να συνειδητοποιούμε τις σφαιρικές επιπτώσεις των επιλογών μας. Οπότε είναι σημαντικό να συζητήσουν οι πρόεδροι των επιτροπών για να έχουμε σύντονισμένη προσέγγιση για αυτό το νομοθέσμα διότι έχει πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Δεύτερο σχόλιο για την νητρορύπανση και την οδηγία. Έχουμε την εντύπωση ότι η αντίσταση, η αρχική αντίσταση σε αυτή την οδηγία ε, ήταν κάτι που τελικά δεν αποφύγαμε και μάλλον ακολουθήσαμε λάθος κατεύθυνση και τελικά δεν μπορούν να αποφύγουν την εφαρμογή της η οδηγή. Ο εισηγητής, νομίζω, κάνει λογικές προτάσεις. Λένε κάποιοι δεν πρέπει να κουμπίσουμε την οδηγία. Εγώ αντίθετα ε, πιστεύω πρέπει να ε, ξεκαθαρίσουμε. Δεν θέλουμε δραστικές αλλαγές. Θέλουμε να διορθώσουμε ένα πρόβλημα της οδηγίας σε σχέση με τη χρήση της ε, ζωικής κόπρου. Υποστηρίζω λοιπόν την κατεύθυνση του ΣΥΓΙΤΗ. Εάν μας ακούν οι γεωργοί, αν και νομίζω ότι ε, καλλιεργούν τα χωράφια τους και βάζουν λοιπάσματα να κάθουν να ακούνε εμάς, αυτό που θέλουν είναι να είναι διαθέσιμα τα προϊόντα λίπανσης να είναι αξιόπιστα και να έχουν καλές οδιές. Ε, για να μπουν μετά οι εισοδιές στην τροφική αλυσίδα και να είναι ασφαλή τα τρόφιμα για τους καταναλωτές αλλά θα ανησυχεί το θέμα τη τιμής. Άρα τα εμπορικά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εμείς ε, ανησυχούμε ήδη για την υπερβολική εξάρτηση από τη Ρωσία για τα ενεργειακά προϊόντα. Τα ή τις ίδιες ανησυχίες θα είχαμε την υπερβολική εξάρτησή μας από για την εισαγωγή λοιπασμάτων, αν αυτή είναι μια επίπτωση των ε, επιλογών που θα κάνουμε. Προσοχή λοιπόν, πώς θα ας σπεύσουμε βραδέως, ας κατανοήσουμε πλήρως όλες τις επιπτώσεις των αποφάσεών μας σε όλες τις επιτροπές και τότε θα μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Είναι σημαντικό για του γεωργούς και το επαναλαμβάνω, παρότι ξέρω ότι μάλλον δεν μας ακούνε αλλά καλλιεργούν ε, τα χωράφια τους, Α φροντίσουμε να είναι θετικές και όχι αρνητικές επιπτώσει. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλέρα. Ναι, Παρόλο που δεν έχουμε αρμοδιότητες για το κάδμιο, βλέπω ότι η συζήτηση έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να αποφαθώ ως προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι άμεσα βιώσιμη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις οριακές τιμές για το κάδμιο. Είναι υπερβολικές αυτές οι οριακές τιμές αποκλείεται να εφαρμοστούν από τώρα. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να μειώσουμε το κάδμιο, αλλά ο χρονικός ορίζοντας και οι οριακές τιμές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αδύνατο να εφαρμοστούν αμέσως. Και πολύ συχνά έχουμε αντίθετες απόψεις ε, με την Επιτροπή ε, περιβάλλοντος. Εδώ είμαι τακτικό μέλος και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, είμαι αναπληρωματικό μέλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι τις απόψεις ε, του, της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σέβομαι εξίσου και τις δύο επιτροπές. Αλλά θεωρώ ότι είναι μη βιώσιμε οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι στιγμή ε, τα φωσφορούχα προέρχονται είτε από τη Ρωσία, ε, τη Φιλανδία και τη Βόρεια Αφρική, το Μαρόκο. Αν ε, θέσουμε τώρα αυτέ τι οριακέ τιμέ, θα δεν θα μπορέσουμε πια να αγοράσουμε ε, φωσφορούχα λιπάσματα από το Μαρόκο. Και δεν το λέω εγώ αυτό, δεν το βγάλα από το μυαλό μου, μας το λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κλάδος και το λένε και όλα τα στοιχεία. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα αποκλείσουμε, αν θεσπίσουμε άμεσα τα νέα, τις νέες οριακές τιμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το κάδμιο, θα αποκλείσουμε το Μαρόκο, θα περιοριστούμε μόνο σε εξάρτηση από τη Ρωσία. Είναι λογική η πρόταση της κυρίας Γκαρντίνη, και σέβομαι τις απόψεις των συναδέλφων, αλλά δεν θα πρέπει να μας ε, έχετε να φέρετε σε αντιπαράθεση να χωρίζετε αυτούς που είναι φιλοπεριβαλλοντικοί, οικολόγοι και όλοι οι υπόλοιποι ε, που δεν ασθενίζονται αυτή τη θέση ότι είναι κατά του περιβάλλοντος. Όχι, ο καθένας έχει τις πληροφορίες του, έχει τη γνώμη του ε, για την κατάσταση και για την απόφαση και δεν είμαι υπέρ των μαξιμαλιστικών θέσεων ούτε εδώ ούτε πουθενά άλλο και δεν θέλω να διαχωρίζετε ε, τους συναδέλφους μεταξύ των φίλων του περιβάλλοντος και των υπολείπων που είναι εχθροί. Ευχαριστώ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, κυρία Γιωχάννα Μπέρτσελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για την Επιτροπή. Θέλουμε ε, να προχωρήσει. Ε, είναι ε, περίπλοκο το θέμα, όπως είπανε πολλοί, ε, από τεχνικής, πολιτικής και νομικής πλευράς είναι στο σταυροδρόμι ανάμεσα σε οδηγία για τα προϊόντα, για τα χημικά, για τα απόβλητα, ε, είναι σε κομβικό σημείο. Εμπλέκονται, όπως και σε εσάς, πολλές ε, υπηρεσίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα μπορώ να κάνω μια προκατακτική ανάλυση ε, από που προκύπτει από τις συζητήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται πιο εφισταμένα με το ζήτημα. Ευχαριστώ πάντως ε, για την ευκαιρία που μου δίνετε για ανταλλαγή απόψε. Ε, έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά για να κατατεθούν αυτές οι υποεξέταση τροπολογίες, το βλέπουμε αυτό. Σε κάποιες από αυτές τις τροπολογίες βλέπουμε νέες ε, ορολογικές έννοιες, ε, ορυκτά, ε, ε, παραδείγματος χάρη λιπάσματα, αντί για ανόργανα λιπάσματα. Ε, βλέπω ότι ε, γίνεται μια προσπάθεια να χρησιμοποιούμε τους όρους της αγοράς ε, για τα λοιπάσματα. Ε, οπότε ναι, να το εξετάσουμε μόλις υιοθετηθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, θέλουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες που μας βοηθήσουν να διερευνήσουμε το, το δυναμικό της ανάκτησης θρεπτικών στοιχείων, διότι αυτό είναι κεντρικό σημείο στην πρωτοβουλία που ανέλαβε και την πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε να θέσουμε εν κινδύνο ούτε τη δημόσια υγεία ούτε το περιβάλλον κάνοντας αυτό φυσικά. Τρεις ανησυχίες ε, μας απασχολούν ε, διαβάζοντας ε, τα σχέδια τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Βιοδιαγέρτες για τα φύτα, πρώτα απ' όλα, για τον ορισμό τους προσοχή τα προϊόντα λίπανσης ε, ε, που θα πρέπει να ρυθμίζονται στον κανονισμό προϊόντων φυτοπροστασίας ε, δεν θα πρέπει να συγχέονται με αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για βιωτικό άγχος για τα φυτά, είναι κάτι που αποκλείεται από, τον, από την οδηγία φυτοπροστασίας και ο στόχος δεν είναι να εκλείψουν από την αγορά τα προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα απλώς ε, υπάγονται στην οδηγία για τα προϊόντα φυτοπροστασίας. Ε, πάλι για τους διδεγερτες πολλές τροπολογίες αποσκοπούν στην ε, νέα μικροβιακού τύπου βιοδιέγερση. Ε, Υπάρχουν προϊόντα που δεν απαριθμούνται στον κατάλογο ε, υπαριθμών 7 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συστατικά στοιχεία και γι' αυτό θέλουμε να είναι πλήρης ο κατάλογος των μικροβιακού τύπου βιδεγερτών στην πρόταση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αναζητείτε την επέκταση του καταλόγου και σε τεχνικό επίπεδο το επεξεργαζόμαστε αυτό το ζήτημα στην Επιτροπή, αλλά για να υπάρχει λογοδοσία είναι σημαντικό ο κατάλογος να αποφασιστεί ή από τους νομοθέτες ή από την Επιτροπή και όχι από οργανισμούς βιομηχανικής τυποποίησης. Όταν ναι, γίνεται διασταυρούμενη αναφορά για τις ενεργές ουσίες των παρασύτοκτων των βιοκτώνων, δεν ε, εξασφαλίζουν αυτόματα το επιθυμούμενο επίπεδο συγγνώμη ασφάλειας, κατά τη γνώμη μας. Δεύτερον, Υπάρχουν προτάσεις για να διαγράψουμε κάποιες διατάξεις του ΡΙΤΣ για την ε, εκτίμηση της ασφάλειας, ε, για χρήση κάποιων προϊόντων. Ε, όταν μιλάμε για χημικά στοιχεία και την χρήση τους και την εκτίμηση της ασφάλειας του ΡΙΤΣ, Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι μιλάμε για πρωτογενείς ε, πρώτες Μόνο ε, για αυτές υπάρχουν εκτιμήσεις, αξιολογίες που προβλέπονται στην πρώτη επιτροπή. Ε, αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει εκτίμηση των κινδύνων. Τέλος, τρίτη παρατήρηση, για την προώθηση της ασφαλούς ανάκτησης θρεπτικών στοιχείων, ε, η πρόταση για την, ε, το περιορισμό των, ε, του, καταλόγου αυτών των λοιπασμών μπορούν να χαρακτηριστούν ως mineral ε, Όταν μιλάμε για οργανικό άνθρακα ή για τη διαλυτότητα του φωσφόρου ή για τον περιορισμό σε ε, κάποιες μορφές ε, υδρογόνου, ε, ε εξετάζουμε το ενδεχόμενο συμπερίληψή του στο μέλλον στον κατάλογο. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει αυτό. Όταν μιλάμε για την αποτελεσματικό και διαθεσιμότητα των φυτών στους γεωργούς, ε, προτείνουμε να γίνει αυτό μέσω της σήμανσης. Αρκεί ε, για το γεωργό ε, να αναφέρονται αυτά τα στοιχεία στη, στην περιγραφή του προϊόντος, στη σήμανση. Υπάρχουν δύσκολες τεχνικές και νομικές πλευρές. Ξέρω και εσείς από πλευρά σας αναλύετε όλα αυτά τα ζητήματα. Είμαστε στη διάθεσή σας και με τα χαράς να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες ε, που θα χρειαστείτε για να καταλήξετε τελικά σε σημαντική λύση στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ εισηγητής ο κύριος Χάιτεμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Πρώτα απ' όλα ακούσαμε πολλά για την οδηγία για την ιτρορύπανση, τα ζωτούχα. Να σας ε, εξηγήσω για ποιου λόγους κατάθεσα τη σχετική τροπολογία. Δεν θέλω να θεωρήσουμε την οδηγία για την ιτρορύπανση. Υπάρχει κάποιο λόγο και θα ήθελα να σα τον πω για να βρούμε λύση από κοινού. Ποιο είναι το διακύβευμα. Σε μερικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο και περισσότερες περιφέρειες αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Εξαιτία τη περιβαλλοντική νομοθεσία, οι γεωργοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, στα χωράφια του όλη την κοπρία που έχουν. Αλλά αντίθετα θα πρέπει να εισάγουν ε, τεχνητά λοιπάσματα, ανόργανα, για να έχουν αρκετέ θρεπτικέ ουσίε για να τροφοδοτήσουν τι καλλιέργειε. Και τι γίνεται με αυτή την κοπριά. Δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στη δική του ε, καλλιέργεια. Θα πρέπει να την εξαγάγουν. Μερικέ φορέ ε, τη χάνει επεξεργασίας και χρησιμοποιείται στο τσιμέντο για την κατασκευή δρόμων και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν αυτή τη παράλληλη κατάσταση. Οι θρεπτικές ουσίες στη ζωική κόπρο να μην χρησιμοποιούνται, να μην αξιοποιούνται στο έπακρο. Και θέλω να λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό. Να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι θρεπτικέ ουσίε από τη ζωική κόπρο με καλύτερο τρόπο, ώστε να μην εξαρτώμαστε από τι θρεπτικέ ουσίε των ε, συνθετικών, των ανόργανων δηλαδή λοιπασμάτων. Και νομίζω ότι η λύση είναι να αλλάξουμε τον ορισμό της ζωικής κόπρου. Δυστυχώς, ο ορισμός αυτός της ζωικής κόπρου περιλαμβάνεται στην οδηγία για την ιτρορύπαση. Εγώ δεν θέλω να αναθεωρήσουμε την οδηγία. Απλώς θέλω να τροποποιήσουμε τον ορισμό της ζωικής κόπρου που ισχύει εδώ και 30 χρόνια, από την οδηγία για τα ζωτούχα, για την μητρολήπαση. Αν δεν αλλάξουμε τον ορισμό για τη ζωική κόπρο, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις θρεπτικές ουσίες της κοπριάς και να κάνουμε ένα λίπασμα με σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που θα αντικαταστήσει το τεχνητό λίπασμα. Αν δεν το κάνουμε όλο και περισσότερο θα χάνουμε τι θρεπτικέ ουσίε από τη ζωική κόπρο γιατί θα μπορεί ο Γιώργο να τις χρησιμοποιήσει στην καλλιέργειά του αυτά φτάσει σε ένα όριο. Αλλά θα είναι υποχρεωμένο, να χρησιμοποιήσει θετικά λοιπάσματα. Ευχαριστώ τον κύριο Ταραμπέλα και θα προσπαθήσουμε και με την κυρία Γκυλέρα να βρούμε μια λύση ώστε να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό της κυκλικής οικονομίας γιατί υστερούμε ως προς αυτό. Και τώρα κάποιε άλλε ανησυχίε που αναφέρατε. Είπατε ότι δεν είναι αρκετά προηγμένη τεχνολογία ώστε να εξάγει ε, τις θρεπτικές ουσίες από τη ζωική κόπρο και να τις αξιοποιήσω καλό λίπασμα. Εγώ διαφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε μια συζήτηση ποιο, είναι, ποιο ήρθε πρώτο, το αυγό ή η κότα. Θέλουμε να συμφωνήσουμε σε κάποια κριτήρια, ώστε να μπορεί ο κόσμος να επενδύει και να έχει τα κριτήρια αυτά ως γνώμονα για να ξέρει προς τα που θα, κατευθυνθεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κριτήρια, δεν υπάρχουν κατευθύνσεις. Οι γεωργοί θέλουν να επενδύσουν αλλά δεν ξέρουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν και έτσι θα αποθαρρυνθούν και δεν θα κάνουν επενδύσεις για να χρησιμοποιήσουν αυτό το δυναμικό. Εγώ θέλω κάποιου ο, κάποιους συγκριτικούς κανόνες, κάποιο γνώμονα και κριτήρια, ώστε στο μέλλον θα είναι έτοιμη η τεχνολογία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και κάποιες νομικές αμφιβολίες τώρα ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον ορισμό για τη ζωική κόπρο στην οδηγία νετρορύπασης μέσω του συγκεκριμένου κανονισμού για τα λοιπάσματα. Εγώ το έλεγξα και μπορούμε να το κάνουμε. Το εξακρίβωσα και μπορούμε να το κάνουμε γιατί το ίδιο κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Αλλάζει τον ορισμό των βιοδιαγερτών, για παράδειγμα, στον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά υλικά. Επίσης, αλλάζει κάποιους ορισμούς για τα υποχόντα ζωικής προέλευσης. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί λοιπόν αυτή η τεχνική να αλλάξουμε τον ορισμό. Ξέρω ότι φοβάστε να αλλάξουμε οτιδήποτε στην οδηγία για τα ζωτούχα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η μόνη λύση, εκτός αν βρούμε κάποια άλλη. Αλλά θα πρέπει με την αλλαγή του ορισμού της ζωικής κόπρου να απελευθερώσουμε το δυναμικό της κυκλικής οικονομίας. Και είπε η κυρία Ντελαέ ότι είναι υποχρεωτικό. Όχι, δεν θα είναι υποχρεωτικό. Απλώς αφήνουμε ανοιχτή αυτή τη δυνατότητα ότι οι θρεπτικέ ουσίε τη ζωική κόπρου που θα πήγαιναν χαμένε ή θα έπρεπε να εξαχθούν ή να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομικό κλάδο να χρησιμοποιηθούν ω πηγή για ένα λείπασμα που θα φέρει το σήμα CE. Θα ήθελα να συνεχίσουμε πάντως τις συζητήσεις, να εμβαθύνουμε για να αναζητήσουμε κοινέ λύσεις και να ε, μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χαίτεμα για τις απαντήσεις σας. Μας έδειξαν και αυτές πόσο σύνθετο και περίπλοκο είναι το πρόβλημα των προϊόντων λίπανσης. Θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε και να συνεννοηθούμε και με τις υπόλοιπες επιτροπές. Εμείς θα ψηφίσουμε εδώ στις 30 Μαΐου την έκθεση Χαίτεμα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σε λίγο θα συνεδριάσουν οι συντονιστές λίγη πρωινή δημόσια συνεδρίαση. Η δημόσια συνεδρίασή μας θα συνεχιστεί το απόγευμα στις 3. Καλό μεσημέρι.